Εδώ έχουμε, ε, ακούσαμε ότι υπάρχει ε, αντιδικαστικό πάλι ε, Κυρία Χάρμσε, κύριε Σούλτς, κύριε Πρόεδρε, για μας πιστεύουμε ότι σε ό,τι αφορά την πρόταση για το μεταβατικό αυτό στάδιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τέσσερις θέσεις πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά και όχι για όλους μαζί. Γιατί? Γιατί η ομάδα μας θεωρεί ότι δεν έχει νόημα καταρχάς για τρεις μήνες μόνο να διορίσουμε καινούργιους επιτρόπους. Αν παρόλα αυτά προχωρήσουμε στον διορισμό επιτρόπων, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο κύριος Oettinger ε, το εξέφρασε αυτό, θεωρούμε ότι θα ήταν σημαντικό μετά τις ακριώσεις ε, τις χθεσινές να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την ψήφο μας για τα διαφορετικά αυτά τέσσερα μέλη. Εμείς δεν θα θέλαμε να καταψηφίσουμε όλους τους υποψηφίους αν μπορούμε να τους ψηφίσουμε ξεχωριστά Εντάξει, γιατί ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα μετά από τις ε, ακροάσεις. Ε, συγκεκριμένα για τον κύριο να αποφανθήκαμε αρνητικά. Σας παρακαλώ αφήστε λοιπόν τους βουλευτές να αποφασίσουν ξεχωριστά. Ιδάλλως θα αναγκαστούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι απόλυτα, απόλυτη ανοησία και για σπατάλη χρημάτων, θα αναγκαστούμε να καταψηφίσουμε ή στην καλύτερη περίπτωση να αποσχούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χάρμς, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Φόξ, κοιτάξτε το λόγο. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Κύριε Φόξ, παρακαλώ, ακούστε με πρώτα. Για το θέμα αυτό ή για άλλο θέμα θέλετε το λόγο για αυτό το θέμα. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Uh, e Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα ECR υποστηρίζει την ε, πρόταση των Πρασίνων. Πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό κάθε υποψήφιος ε, να ε, αντιμετωπίζεται επί της αξίας του και υπάρχει ένας υποψήφιος τον οποίο δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε και άρα θα αναγκαστούμε λόγω της δικής σας απόφασης να καταψηφίσουμε και τους τέσσερις. Και είναι σημαντικό τα μέλη να γνωρίζουν τις οικονομικές συνέπειες αυτής της ψήφου. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι ορίζοντας αυτούς τους τέσσερις τέσσερις προσωρινούς επίτροπους θα λαμβάνουν τα ωφέλη του ότι τέλεσαν επίτροποι για το υπόλοιπο της ζωής τους παρότι έχουν θητεύσει μόνο τρεις μήνες. Die, also η τελευταία ερώτηση είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Θα πρέπει να τα κοιτάξω. Δεν, δεν, ξέρω τι γίνεται για το υπόλοιπο τη ζωή του δηλαδή. Καλό, καλό και όμορφο θα ήταν. <laughs> Θα ενημερωθώ, λέει ο πρόεδρο. ich weiß überhaupt nicht, warum Sie δεν ξέρω γιατί είστε τόσο νευρικοί όταν δεν ε, λαμβάνετε απάντηση φωνάσατε πριν ε, ακούσατε καν τι έχω να πω. Εκπληκτικό. Λοιπόν, καταρχά η διάσκεψη των Προέδρων διαπίστωσε ότι η ψηφοφορία αυτή θα πρέπει να γίνει συνολικά, unblock. Ε, αυτό το ψηφίσαμε χθε στην διάσκεψη των Προέδρων και η σαφή πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ τη συνολική ε, ψηφοφορία. Η κυρία Χάρμσε λοιπόν έκανε αίτημα για να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Ένα υπέρ, ο κύριο Φόξ, θέλει να μιλήσει και κάποιο κατά, ο κύριο Σάια. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Επειδή έχουμε και άλλη μία ψηφοφορία ενώπιόν μας για το καινούριο σώμα των επιτρόπων. Θα ψηφίσουμε λοιπόν unblock ε, συνολικά σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία αυτή και αυτό ακολουθεί τους ε, κανόνες που ισχύουν για την ψηφοφορία της Επιτροπής. Και εκεί θα ζητήσετε λοιπόν ξεχωριστές ψηφοφορίες. Τι θα κάνετε. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να κάτσουμε να ξαναγράφουμε συνέχεια τις παλιές και τις πρώτερες αποφάσεις γιατί αλλάζουν γνώμη οι συνάδελφοι. Στις επιτροπές παρόλα αυτά υπήρχαν ευκαιρίες αυτές και ε, φέρατε λοιπόν και χρησιμοποίησατε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, την δυνατότητα να ψηφίσετε ξεχωριστά, να καταψηφίσετε και χάσατε. Τι θέλετε να ξαναχάσετε και εδώ, εμεί δεν υποστηρίζουμε αυτό το αίτημα. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο. Κυρίε και κύριοι, κυρία Τσίμερ, δεν θα ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση. Έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ για διαδικαστικό μόνο. Ναι, να ανοίξτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ένα διαδικαστικό θέλω να θέσω κι εγώ. Θα ήθελα να ξέρω αν για την, ε, το διορισμό, τον δεύτερο διορισμό έτσι, επιτρόπων είναι υποχρεωτικό να ψηφίζουμε unblock, γιατί δεν πρόκειται για διορισμό όλου του σώματος των επιτρόπων. Εγώ δεν γνωρίζω και για την μετέπειτα διορισμό επιτρόπου να ισχύει αυτός ο κανόνας για την συνολική ομαδική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Τσίμερ, η ψηφοφορία η ομαδική συνολική unblock δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι να ψηφίσετε συνολικά η καινούργια επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τους μετέπειτα διορισμούς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Αυτό υπόκειται στην ευχέρεια του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό λοιπόν χθες στην διάσκεψη των Προέδρων που ήσασταν κι εσείς έθεσα το θέμα και εκεί διαπίστωσα και όχι μόνο εγώ αλλά και οι υπόλοιποι διαπίστωσαν γιατί δεν είναι δική μου η απόφαση δεν είναι μόνο δική μου η απόφαση. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η διάσκεψη των Προέδρων υπήρχε ευρία πλειοψηφία για να ψηφιστούν συνολικά αυτοί οι τέσσερις ε, ε Λοιπόν, η κυρία Χάρμς ζήτησε λοιπόν να διορθωθεί αυτή η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων και να ψηφίσουμε και νομίζω ότι είναι δίκαιο να ψηφιστεί η πρόταση της κυρίας Χάρμς. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Χάρμς. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται το αίτημα. τώρα λοιπόν περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία για τους τέσσερις επιτρόπους. μπλοκ. Όλοι μαζί. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο Το Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχει τις ε, χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός νομοθετικού κειμένου. Σας ερωτώ λοιπόν, ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες της εκλογής των τεσσάρων επιτρόπων για τρεις μήνες. Τουλάχιστον θα πρέπει να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι αυτή την πληροφορία πρέπει να την έχουμε πριν ψηφίσουμε. Diese οι επίτροποι αυτοί εκλέγονται για το υπόλοιπο της θητείας. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου η επόμενη θητεία θα ξεκινήσει και θα αναλάβει τα καθήκοντά της από 1η Νοεμβρίου. Υποψήφοι λοιπόν που θα ψηφίσουμε τώρα ξεκινούν τώρα άμεσα τη θητεία τους και θα λήξει η θητεία τους στις 31 Οκτωβρίου. Καθίστε, δεν έχω τελειώσει ακόμα, λέει ο πρόεδρος. Ίσως να περιμένετε να τελειώσω τι ευγενική που είσαστε. Ευχαριστώ. Τώρα, τώρα όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα επιδόματα, θα γνωρίζετε ότι αυτά προκύπτουν από τους κανονισμούς για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία οι κανονισμοί αυτοί διατίθενται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συνταξιοδοτικά προβλέπονται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο website και του Κοινοβουλίου. Να περάσουμε στην ψηφοφορία τώρα. Αν δεν τα γνωρίζετε αυτά, κύριε Λούκε, να μην δίνετε την εντύπωση ότι είστε τέλεια ενημερωμένος. Όχι, τώρα θα ψηφίσουμε τα τέσσερα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους υποψηφίους, έναρξη ονομαστικής κλίσης. Αν όλοι ψήφισαν, πέρασε της υποφορίας. 421 ψήφοι υπέρ, 170 κατά, 32 αποχές, οι τέσσερις ε, λοιπόν ε, επίτροποι εγκρίνονται και διορίζονται. Μάλιστα λοιπόν κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε δήλωση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων και το λόγο έχει ο Επίτροπος.

Good morning, colleagues. Καλημέρα σας συνάδελφοι. Καλημέρα συνάδελφοι. Παρακαλώ όσοι παραμένετε για τη συζήτηση θέλουμε να ξεκινήσουμε. Όσοι αποχωρούν παρακαλώ να αποχωρήσουν γρήγορα, γρήγορα και ησύχως. Θα ξεκινήσουμε με ορισμένες ανακοινώσεις. Please colleagues, could you clear the chamber? Παρακαλώ, αποχωρήστε ησύχω όσοι θέλετε να φύγετε, παρακαλώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάποιες ανακοινώσεις. Ε, οι αρμόδιες ισπανικές αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Χαβιέρ Κόουσο, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Βίλι Μέγερ από τις 15 Ιουλίου 2014. Παρακαλώ. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Είχατε έναν άκρο πεπειραμένο πρόεδρο στο πρώτο τμήμα της Συνόδου και τώρα έχετε μία πολύ άπειρη πρόεδρο στο βήμα. Σας παρακαλώ λοιπόν δείξτε λίγη επίοικια στην απειρία μου. Πάντως θα είμαι σκληρή, σας προειδοποιώ. Συνεχίζω λοιπόν και παρακαλώ να με προσέξετε για μια τελευταία φορά το λέω. Βλέπω ότι εξακολουθούν να συνομιλούν κάποιοι συνάδελφοι. Εγώ συνεχίζω πάντως δυνάμει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης ε, περιεκλογής ε, των ε, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και άρθρο 4 παραγραφο 1 1-4 του κανονισμού σημειώνει το Κοινοβούλιο την εκλογή του κυρίου Χαβιέρ Κάουσο Σοπερμούη με ισχύ από την 15η Ιουλίου 2014. Καλωσορίζω τον νέο συνάδελφο και αναφέρω ότι δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού μέχρι να ε, αληθευτούν τα διαπιστευτήριά του και να δούμε ε, αν υπάρχουν ενστάσεις ε, ε, θα ε, συμμετέχει ως βουλευτής στο Κοινοβούλιο και στα όργανα με πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του με την προϋπόθεση ότι έχει ε, υποβάλει προηγουμένως τη δήλωση ότι δεν ασκεί κάποιο μη συμβατό με την έδρα του βουλευτή καθήκον. Επίσης η ομάδα του ΕΛΚ ζητά τροποποίηση κάποιων μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κατάλογος των ορισμών θα περιληφθεί στα πρακτικά και αν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι την έγκριση των πρακτικών, θεωρούνται αυτές οι τροποποίησεις και ορισμοί ότι εγκρίνονται. Πέρα των ανακοινώσεων και περνάμε στην έναρξη της σημερινής συζήτησης. Παρακαλώ εκ